για τις ψηφοφορίες. Άμα μας βοηθήσετε θα τα πετύχουμε σε πιο γρήγορα. Να κοιτάξουμε τις αντιπροσωπίες για το σχέσεις με το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο. Ποιος είναι υπέρ. Μία ψηφοφορία είναι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Φερέιρα. Ονομαστική κλίση. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Άλλη μια εκθέση Φερέρα. Πάλι με ονομαστική κλίση. Έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Φαντάλων για την ε, αλευτική σύμπραξη. Ονομαστική κλίση, έναρξη ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Άλλη έκθεση Φαντάλεν σε ό,τι αφορά το πράσινο κροτήριο αυτή τη φορά. Ονομαστική κλίση. Έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παραγράφος 4 του αρχικού κειμένου σε τρία τμήματα. Έτσι αυτό καταπιπτεί το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφιστε παρακαλώ όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Περάω Σάντος. Σεράου Σάντο, ε, αλευτική σύμπραξη με τη Μαγαδασκάρη, ονομαστική κλίση, έναρξη πληροφορία. Ούτε εσεί ε, μπορείτε πιο γρήγορα, ούτε οι τεχνικοί μπορούν πιο γρήγορα. Σα παρακαλώ. Τώρα ψηφίζουμε. Ψηφίζονται όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Σάλμπα Μπιντεγκάιν, πρωτοκόλλα για την τροποποίηση τη Συμφωνία του Μαρακέ για την ιδρύση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Και για τι δύο εκθέσει ε, ο εισηγητή ζήτησε δύο λεπτά. Ο κύριος Ζάλμπα Μπιντεγκάιν έχει το λόγο. Πάρα πολύ σύντομος θα, είμαι. Ε, θέλω να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλειά αυτή που έγινε με την έκθεση. Είναι μια συμβολή στο παγκόσμιο εμπόριο, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και λόγω της ε, πρόκλησης της μετανάστευσης που αντιμετωπίζουμε αν κατορθώσουμε να βρούμε μία λύση στην πηγή του προβλήματος νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιου είδους εργαλεία έτσι ώστε να προάγεται η οικονομική ανάκαμψη σε χώρους όπου είναι κυρίως απαραίτητη. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι, είναι ονομαστική κλίση για την πρώτη έκθεση. τη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερη έκθεση για τα παιδικά σχεδόν ταυτόσιμο για τις ε, διευκόλυνση του εμπορίου. 11, τροπολογία 11, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Οι 2 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Οι 12 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. η 13 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Η 3 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Η 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 4. Έναρξη ηλεκτρονική ψηφορία. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 8 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται η 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση παρακαλώ ένας ψηφορίας ψήφισατε όλοι πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνετε. και τώρα πάμε στην ε, έκθεση Σβόμποντα εξουσιοδότηση Αυστρίας, Βελγίου και Πολωνίας για τη σύμβαση ε, για τη συμβάση των πραγματικών μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών Ονομαστική κλίση, παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην έκθεση της κυρίας Κέλλη για τα προσωρινά στον τομέα της διεθνής προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα. Έχουμε κάμποσες τροπολογίες όλες μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 27 έναξη ψηφορίας παρακαλώ ηλεκτρονικά. Εάν ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Έχουμε προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχουμε προφορική τροπολογία εδώ που συμφωνήθηκε από του Κιώδη. Είναι μια ενημέρωση σε σχέση με αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί για τι νέε προτάσει του Γιούγκερ. Έχετε λοιπόν στον καταλογό ψηφοφορία επειδή είναι δύσκολο να διαβάσετε, αλλά αυτό που λέμε είναι ότι μία περαιτέρω με την κατάσταση 120.000 ατόμων από την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα θα περιληφθεί στη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό λέει η πρόταση και θα το βρείτε στον κατάλογο τη ψηφοφορία για να μην σα τα διαβάσω και είναι περίπλοκα τα πράγματα. Ευχαριστώ, λέει κυρία, ο πρόεδρο, κυρία Κέλλερ. Υπάρχουν αντιρρήσει, παρακαλώ. Είναι πιο πολύ από 40 οι βουλευτέ που σηκώθηκαν. Θα ψηφίσουμε στην αρχική μορφή λοιπόν την ε, τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ για την 47 στην αρχική της μορφή παρακαλώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε παρακαλώ όλο. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 29 καταπίπτει, 44 στα δύο τμήματα, πρώτο τμήμα με, ονομαστική κλίση. Haben alle abgestimmt? Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 34 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Έλεγχος. Ζητείτε για την 48. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναξη ψηφοφορίας. Εάν ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 42 με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Έναξη ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 43. Με ονομαστική κλίση. Έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 3. Με ονομαστική κλίση. Έναρξη ψηφοφορία. Εάν ψήφισατε όλοι. ολοκληρώνονται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η τέσσερα με ονομαστική κλίση. Έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Έλεγχο για το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, τη 5. Ένα ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 6 με ονομαστική κλίση, παρακαλώ, Ένα ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και 45 καταπίπτει αυτού του. Η 9 με ονομαστική κλίση παρακαλώ έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 46 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Έλα, έχουμε την 46 παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 13 με ονομαστική κλίση, παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε και άλλες ε, ονομαστικές κλήσεις. 14. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 15. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 16. Έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται η 18. Έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται η 19. Έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 22. Έναξη ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 23 παρακαλώ ένα ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα, παρακαλώ. Με ονομαστική κλίση. Άλλαξη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην έκθεση Westphal για την αστική διάσταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξεκινήσουμε με την παράγραφο 20 με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Ένα ψηφοφορίας. Ψήφισετε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 26 σε δύο τμήματα παρακαλώ το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ε, με ονομαστική κλίση ένα ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, άνοιξη ψηφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα το ψήφισμα όπω τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορίας, παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην έκθεση Τάματόιτς για τι επενδύσει για θέσει εργασία και ανάπτυξη. Προώθηση τη οικονομική, κοινωνική και ταυτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξεκινάμε στην παράγραφο 4 του αρχικού κειμένου, σε δύο τμήματα παρακαλώ, με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα, έναρξη ψηφορία. Ψήφισετε όλοι παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη ψηφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 22 του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 24 του αρχικού κειμένου ε, ονομαστική κλίση έναρξη. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 24 σε 27 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορίας. Εάν ψηφίσατε όλοι, ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Ψηφίσατε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παραγράφος 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 29 σε δύο τμήματα επίσης με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα παρακαλώ ανεξιψηφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, Ένα ψηφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παράγραφος 30. Σε τρία τμήματα με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα, παρακαλώ. Ψήφισετε. Ψήφισατε όλοι, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία λοιπόν. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται τρίτο τμήμα, παρακαλώ. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται Παράγραφο 45. Ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται παράγραφο 64 σε δύο τμήματα πάντα και τα δύο με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 66 σε δύο τμήματα με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Αν ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη ψηφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος έναξη ψηφοφορίας. Να ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε... Στην έκθεση βάντακα. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, ε, πέρασα ένα φίλο, έχουμε την έκθεση Κούκαν προηγουμένως για το 2012 για την ενεργή γύρανση το έτος αυτό και την αλλαγή μεταξύ γενναίων. Ψηφίζουμε ε, ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ στην παράγραφο 8 κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17 σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο υπέρ Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18 σε δύο τμήματα. Το τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 28 υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται. Παράγραφος 30 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 39 σε τρία τμήματα, τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά, Άποχες. Υποθέτω ότι εγκρίνεται, αλλά μάλλον ε, χρειάζεται επαλήθευση. Αρχίζει τώρα αυτή τη στιγμή ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην έκθεση Βαντεκάμπ με θέμα την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές το 2011. Παράγραφος 3. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 4 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. Ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 11 ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Εάν ψηφίσατε όλοι, πέρας, εγκρίνεται. Παράγραφος 13 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέ. κατά, αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 16 ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Εάν ψηφίσατε όλοι, πέρας, angenommen. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο ονομαστική ψηφοφορία άρχεται τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγράφος 20 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 26. Ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Εάν ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 29. Ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34. τι παύλα. Παρακαλώ αρχίζει η ψηφοφορία με ηλεκτρονική επαλήθευση και ονομαστική κλίση. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34. Η 12η παύλα σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 41 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 43 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφος 54 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφος 60 σε δύο τμήματα υπέρ του πρώτου, κατά εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά εγκρίνεται. Παράγραφος 63, Παύλα 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 πάντα, Παύλα 5, σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ονομαστικά, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πάντα στην παράγραφο 63, Παύλο 8, ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 63 είναι ένα τη Παύλα σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη ονομαστική είναι αυτή η ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα. Και αν ψηφίσατε όλοι. Κλείνει. Εγκρίνεται. Παράγραφος 63, δέκατη παύλα, ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 63, δωδέκατη παύλα, ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 64, Παράγραφος 64, Παύλα 5, υπέρ. Πέμπτη, Παύλα, ειπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η έβδομη, Παύλα, πάντα στην 64, είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η εντέκατη, είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και πάντα στην 64, 12η Παύλα, σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 παύλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα είμαστε στην παράγραφο 65 πρώτη παύλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η πέμπτη παύλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η έκτη ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη 12η Παύλα σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 66, 8η Παύλα, υπέρ, κατά, κατά. Ξανά, υπέρ, δεν σας βλέπω. Κατά. Υποθέτω ότι έχει απορριφθεί, αλλά χρειάζεται απολύθευση. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική απολύθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφο 66, ένατη παύλα, σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη G σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα του ψηφίσματο με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Εάν ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση της κυρία Βόζεμπεργκ στα διαδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο. Έχουμε την παράγραφο 22. Παράγραφος 22, το αρχικό κείμενο ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Είναι η έκθεση της κυρίας Βόζεμπεργκ, παράγραφος 22. Αρχίζει η ψηφοφορία ονομαστικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. παράγραφος ονομαστικά και πάλι αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 35 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ε, πέρασε. Εγκρίνεται. Η 42 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφο 48 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη R, λατινικό, ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα. Και αν ψηφίσατε όλοι, λίγοι. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, ακολουθεί έκθεση Ροντρίγκε με θέμα την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της εκπαίδευσης έχουμε λάβει από την e ΕΝΕΦ την ε, ε, ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για ένα εναλλακτικό ψήφισμα. Το αρχικό κείμενο λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της παραγραφού 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 5 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο. Θέλετε έλεγχο. Ωραία. Το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 1 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Τι θέλετε. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 5. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, παράγραφος 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 21 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 27 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 28 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 29. Σε τρία τμήματα πάντα ονομαστικά. Πρώτο τμήμα αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Αν ψηφίσατε όλοι. Καλό θα ήταν και το ΕΛΚ να μου κάνει κανένα νόημα να ξέρω πώς ψηφίζει. Πώς να ψηφίσω εγώ δηλαδή. Ε, ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Πάλι ονομαστικά αρχιτή ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 30 ονομαστικά, αρχιδή ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 31 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 40 υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγουσα 41 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 ε, σε τρία τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το τρίτο υπέρ έλεγχο ζητάτε για το 2. Αρχίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά να επαληθεύσουμε το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Το τρίτο τώρα τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 49 σε τρία τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το τρίτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 50 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον υπέ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπε κατά, αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 53, δύο τμήματα και πάλι, τμήμα πρώτο υπέ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη G σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη έρθει σε δύο τμήμα, τσεκ φωνές από κάτω. Ωραία. Ελέγχουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα της G, αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη T ΤΑΦ ε, υπέρ. Τι ήταν αυτό, το δεύτερο τμήμα, δεν ήταν τη ΕΡ. It was Ζητώ συγγνώμη. Η σκέψη ΕΡ σε δύο τμήματα. Το τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα είναι το τι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. So, wir kommen zum letzten... Και έχουμε την τελευταία έκθεση τώρα, έκθεση ΣΦΑΠ, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Ελβετία. Εμπόδιο όσο αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς είναι μία και μόνη ερμαστική ψηφοφορία. Αφήστε τις κάρτες σας παρακαλώ μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Καλή σας όρεξη και ευλογημένη.